Good afternoon everybody Καλό απόγευμα σε όλους. Παρακαλώ καθίστε. Για να ξεκινήσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, η ψηφοφορία θα κρατήσει περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Ε, εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να υιοθετήσουμε την ε, ημερήσια διάταξη, σημείο 2, σημείο 3 τα πρακτικά της συνεδρία τη 23 η και 24 η Ιανουαρίου έχουν διανεμηθεί σε όλα ε, τα μέλη της Επιτροπής μας. Εάν δεν υπάρχουν ε, θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκαν. Έχω κάποιες ανακοινώσει. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Και έχω μια μεγάλη σειρά αποφάσεων των συντονιστών που θέλω να διατρέξω μαζί σας έγκριση της ημερήσιας διάταξης, όλα ε, όσα ζητήθηκαν ε, έγιναν δεκτά. Δεν χρειάζεται να σας τα διαβάσω όλα, ρωτήστε το συντονιστή σας. Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις, η έκθεση για την πρωτοβουλία πολιτών ε, θα γίνει από την Άλντε. Η νομοθετική έκθεση πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας πολιτών ε, θα την αναλάβει το ΕΛΚ. Θα είμαστε συνδεδεμένοι σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού ε, και η επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή θα είναι η ΑΦΚΟ. Ε, συστάσεις. Εξετάσαμε τα θέματα αυτά όσον αφορά το Brexit. Έχουμε λάβει 120 αναφορές λόγω της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ψηφίστηκαν και θα γίνει μια κοινή ακρόαση ΛΥΜΠΕ, ΕΜΠΛ και ΠΕΤΗ κάποια στιγμή την Άνοιξη, Απρίλιο, Μάιο ή Ιούνιο φέτος αποφασίσαμε σχετικά με τι διερευνητικέ επισκέψεις θα πραγματοποιηθεί μία ήδη τον Μάιο στην Ισπανία, πριν το καλοκαίρι δηλαδή, με πέντε μέλη και τέσσερα εξοφίσιο μέλη. Και συζητήσαμε και τι διερευνητικέ επισκέψεις για το δεύτερο μισό του 2017, για το δεύτερο εξάμεινο. Το δίκτυο ΠΕΤΗ θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ήδη τον Μάρτιο. 21 Μαρτίου στις 2 η ώρα το απόγευμα. Πρόκειται για μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Και καλούμε όλη την Επιτροπή να συμμετάσχει στο θέμα αυτό. Ομάδα εργασίας ε, για την ε, ευμερία των παιδιών, ε, όπου προεδρεύει η Ελεονόρα Εύη, ολοκληρώνει τις εργασίες της ολοκληρώνει το έγγραφο με βάση τη συμβολή διαφόρων εμπειρογνωμόνων και θα μπορέσουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας να ψηφίσουμε πάνω στις συστάσεις. Όταν γίνει αυτό θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της η ομάδα εργασίας για την ευημερία των παιδιών. Τι άλλο έχω να σας πω. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων ε, σχετικά με τις ε, ε, παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ολομέλεια κατά την υπερψήφιση της ε, έκθεσης και αποφασίστηκε να στείλουμε επιστολή στον Πρόεδρο Ταγιάννη όπου να αναφέρουμε τι έγινε κατά διάρκεια της συνεδρίασης, να περιγράφουμε την κατάσταση. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω ε, σχετικά με την συνεδρίαση των συντονιστών και έτσι προχωράμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης, ψηφοφορία. Σας παρακαλώ λοιπόν τοποθετήστε τις κάρτες σας ε, στις συσκευέ. Και ας ελέγξουμε, να δούμε καταρχάς, ε, να διαπιστώσουμε καταρχάς αν είμαστε όλοι παρόντες έναρξη της ψηφοφορίας ε, για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε αρκετά μέλη από κάθε ομάδα. Έχουμε τη σωστή αναλογία μεταξύ των ομάδων. Από ό,τι φαίνεται μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Σχέδιο ψηφίσματος ε, για σύντομο ε, ε, τροπολογία, ε, ε, αιτιολογική σκέψη Β. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση αμέσως. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F. Ε, κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, τμήμα 4. Υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τμήμα 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη G. Πάλι κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ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 Διαγραφή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με τα κατατμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη J σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη K υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη L υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση του δεύτερου τμήματος έναρξης ψηφοφορίας για το δεύτερο τμήμα. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφο σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Παράγραφος 4. Υπέρ. Για την διαγραφή μιλάμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κατόπιν έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το πέμπτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έκτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Παραγράφος 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11. Προφορική γλωσσική φύση τροπολογία ψηφίζουμε. Όχι. Είναι γλωσσική φύση. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα. Απορρίπτεται κατά μία ψήφο. Παράγραφος 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε. Έναρξη της ψηφοφορία. για το δεύτερο τμήμα. Απορρίπτεται. Παράγραφος 17. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παραγράφος 19 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Συγγνώμη, το τμήμα της διαγραφής υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Παράγραφος 22. Προφορική γλωσσική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα ψηφοφορία, το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας πάνω στο δεύτερο τμήμα. Η λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά μία ψήφο αυτή τη φορά. Και το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, το έγγραφο στο σύνολό του, έναρξης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συγχαρητήρια σε μένα λοιπόν. Και ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. So, I'm opening the vote. Ξεκινώ την ψηφοφορία. Όχι. Ξεκινώ τη συζήτηση περί της ε, γνωμοδότησης για το Βρυξέλλες 2α και πρώτα απ' όλα ο εισηγητής. Η εισηγήτρια είναι η κυρία Καμπεσόν Ρουής, την οποία αντικαθιστά η κυρία Ροζιέρ. Σας δίνω λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πράγματι εκπροσωπώ εδώ τη συναδελφό Καμπεσόν Ασολεδάτη που δεν μπορούσε να είναι εδώ ε, σχέδιο έκθεσης που αφορά μια πρόταση αναδιατύπωσης ε, του κανονισμού ε, Βρυξέλλες 2α που καθιερώνει τους κανόνες συνεργασίας σε θέματα οικογενειακού δικαίου ώστε να αναπτυχθεί ένας χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων βασισμένος στην αμοιβή εμπιστοσύνη άροντας τα εμπόδια που εμποδίζουν την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων ε, με τρόπο ικανοποιητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και φυσικά με στόχο την βέλτιστη προστασία των συμφερόντων του παιδιού ε, απλουστεύοντας τις διαδικασίες αλλά και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ πρόκειται για μια διαδικασία διαβούλευσης οπότε η, γνώμη του, η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου δεν δεσμεύει το Συμβούλιο. Δεδομένου αυτού, οι τροπολογίε που προτείνει η συναδελφό μου στο σχέδιο γνωμοδότησή τη αφορούν τα ακόλουθα σημεία. Το πρώτο αφορά το ζήτημα των σεξιστικής φύσης παραβιάσεων κατά του ατόμου λόγω δηλαδή φίλου κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Δεύτερη πτυχή αφορά την ακρόαση του παιδιού. Ουσιαστικά οι μαρτυρίε των παιδιών πρέπει να αποτελούν ένα από του σημαντικότερου παράγοντε που θα λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων, επειδή τα παιδιά είναι το αδύναμο παράγοντα στη διαδικασία αυτή, οπότε τα δικαιώματά του πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο σεβασμού. Ε, τρίτη πτυχή, η διαμεσολάβηση να διευκολύνεται μεταξύ των γονέων κάθε φορά που αυτό είναι δυνατόν. Επίση πρέπει να αναφέρεται ότι οι ακροάσει των παιδιών πρέπει να γινόνται με τη βοήθεια επαγγελματιών και ψυχολόγων διότι πρόκειται για καταστάσεις ιδιαίτερα δύσκολε για τα παιδιά οι περιπτώσει αυτέ της σε θέματα οικογενειακού δικαίου ώστε να εξομαλύνεται η σχέση μεταξύ παιδιού και γονέων σε περιπτώσει δύσκολε, Τέταρτο σημείο. Ακόμα και η οικονομική κατάσταση ενός γονέα είναι σημαντικός παράγοντας, δεν πρέπει να είναι καθοριστικός στην αξιολόγηση τη ικανότητα ενό γονέα να ασχοληθεί με το παιδί του. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλε παράμετροι. Πέμπτο σημείο, να ενισχυθεί και η ενημέρωση των γονέων σε όλη τη διαδικασία, να είναι πλήρη η ενημέρωση στη γλώσσα των λογότομων. Και τελευταίο σημείο, όπω συχνά εκφράζεται αυτή η επιθυμία, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση της αναδιατύπωσης πέντε χρόνια μετά τη θέση ισχύ της. Αυτά είναι τα πέντε βασικά σημεία στο σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Καμπεσόν και αναμένω να ακούσω παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ και δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ECR θεωρεί σημαντική την ε, το σχέδιο της γνωμοδότησης, το οποίο έχουμε να συζητήσουμε, όπως είπαμε αφορά την ε, αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων που έχουν σχέση με τις γαμικές διαφορές επίσης τις διαφορές της γονικής μέρημνας, αλλά και θέματα που έχουν σχέση με την διεθνή απαγωγή παιδιών. Είναι γνωστό ότι στη φάση που επικρατεί πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων έχουμε πάρα πολλούς μικτούς γάμους, αλλά βεβαίως έχουμε επίσης και τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως ε, έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες λύνουν το γάμο ε, οι οποίες βεβαίως πρέπει να εκτελούνται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Πολύ δε περισσότερο έχουμε αποφάσεις που αφορούν την γονική μέρημνα των τέκνων. Έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις αν θέλετε σε πολλά κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει πολλές φορές και αδυναμία της εκτέλεσης αυτών των αποφάσεων. Πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, και παραβιάσεις από την πλευρά ενός εκ των γονέων. Ε, γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή η ρύθμιση η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Νομίζω ότι το βασικό θέμα που πρέπει να μας πασχολεί είναι το ίδιο το συμφέρον του παιδιού. Αυτό είναι ο βασικός πυρήνας γύρω από τον οποίο πρέπει να αρθρωθεί η νομοθεσία. Και εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σημαντικά την θέληση του ίδιου του παιδιού διότι δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες ε, είναι ε, αντίθετες με τη θέληση του παιδιού. Ιδίως δε όταν το παιδί έχει μια ηλικία μεγάλη. Είτε αν είναι 13 ετών και άνω, που σημαίνει ότι έχει δυνατότητα να πει την άποψή του και βεβαίως θα πρέπει αυτή η άποψη να την υπόψη και στις τροπολογίε που βλέπω υπάρχει και η άποψη ότι τα παιδιά τα οποία είναι από 16 ετών και άνω, εφόσον εκφράσουν σχετική επιθυμία, αυτή η επιθυμία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και από τα δικαστήρια. Επομένως θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η νομοθεσία πρέπει να παρέμβουμε στα σημεία που είδαμε ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σωστά στα κράτη-μέλη ή επίσης έχει αναδείξει πολλά προβλήματα, να βελτιώσουμε με τροπολογίες αυτή την νομοθεσία, με πυρήνα βεβαίως κυρίως την, το συμφέρον του ίδιου του παιδιού, με στόχο επίσης να ε, χτυπηθεί η βία η ενδοοικογενειακή που αναπτύσσεται και να υπάρχει φυσικά ίση μεταχείριση των φύλων ε, στις περιπτώσεις εφαρμογής της νομοθεσίας. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία εμείς θέλουμε να θίξουμε και θα έχουμε την ευκαιρία και με τροπολογίες αλλά και στην πορεία να βελτιώσουμε σε συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους συναδέλφους το κείμενο το οποίο θα εγκριθεί από την ε, Επιτροπή μας λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως ότι η ακρόαση του παιδιού είναι ένα σημαντικό δικαίωμα που προβλέπεται από το άρθρο 24 παράγραφος 1 του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το άρθρο 12 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. On this matter. Και εγώ σας ευχαριστώ, δίνω το λόγο σε εσάς κύριε Εύη επί του θέματος. Ευχαριστώ πρόεδρε, λοιπόν, ως δεδηλωμένο στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση αναδιοτύπωση του Βρυξέλλε 2α είναι να εξελιχθεί περαιτέρω ο Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνη και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων βάσει τη αμοιβαία εμπιστοσύνη, εξαλείφοντα τα εμπόδια που ε, αποτελούν πρόσκομα για την ελεύθερη κυκλοφορία. Στην περίπτωση των δικαστικών αποφάσεων, προστατεύοντας καλύτερα τα συμφέροντα του παιδιού. Η πρόταση εμφανίζεται βάσει της αναθεώρησης του προγράμματος, ε, βάσει του προγράμματος REFIT. Βασίζεται και στη δημόσια διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν πολλοί ενδιαφερόμενοι και την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή και όπου διαπιστώθηκαν διάφορα κενά όσον αφορά την γονική ευθύνη. Θεωρήθηκε ε, σωστό να γίνουν κάποιες διορθώσεις ε, στις οποίες θα επικεντρωθούν οι τροποποιήσεις. Στα συμπεράσματα η Επιτροπή καταλήγει να λέει ότι επειδή η δικαστική συνεργασία και η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών έχουν πλέον οριμάσει αρκετά, είναι δυνατόν να περάσουμε σε ένα σύστημα κυκλοφορίας των αποφάσεων πιο απλό και λιγότερο δαπανιερό. Ε, εξαλείφοντας τις διατυπώσεις που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Μετά από αυτή τη σύνοψη και πέραν όλων των ε, όμορφων δηλώσεων ε, της Κομισιόν για τους στόχους που πρέπει να επιδιώξουμε, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, να πούμε τα πράγματα όπως έχουν και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, πώ ασκείται πραγματικά η δικαιοσύνη όσον αφορά το οικογενειακό δίκαιο στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι επί του θέματο η Ένωση έχει μόνο ε, συναρμοδιότητα με τα κράτη-μέλη όπου οι στόχοι που σχετίζονται με την αναδιατύπωση υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν από ορισμένα κράτη-μέλη, από ορισμένα από αυτά, πιο συγκεκριμένα από όσους ε, συγκεκριμένα θέλουν να κινηθούν προς την αντίθετη κατεύθυνση όσον αφορά τα αποτελέσματα και έτσι επιμένουν σε διαδικασίες, σε πρακτικές ε, σε μηχανισμούς που έχουν οδηγήσει σε πολλές καταγγελίες στη δική μας Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, αυτή η ελλειπής εστίαση σε αυτή την πτυχή θα οδηγήσει ε, σε αδιέξοδο όποιε πρωτοβουλίε και να λάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε σε αυτήν εδώ την επιτροπή μα πρέπει να πούμε όπου τόσοι πολλοί πολίτες έχουν στραφεί με τις αναφορές ε, δηλώνοντας σοβαρότητες παραβιάσεις των θεμελιδών δικαιωμάτων που θέλει να διορθώσει ε, αυτή εδώ η αναδιατύπωση οδηγηθήκαμε να δημιουργήσουμε και μια ομάδα εργασίας της οποίας την προεδρία έχω εγώ, έχω την τιμή να προεδρεύω εγώ και δεδομένης ε, και της αδιαφάνειας που συνεχίζει όσον αφορά τις ε, διάφορες τους ε, αμφισβητούμενους μηχανισμούς και πρακτικές των κρατών μελών και λόγω και της μη διαθεσιμότητας των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών που καλούνται να ε, δώσουν αναφορά και να λάβουν τις ευθύνες τους και να συνεργαστούν. Αναφέρομαι για παράδειγμα μεταξύ πολλών, να δώσω το παράδειγμα των γερμανικών αρχών του Jugendamt, του Γραφείου Νεολαίας που συμμετείχε στην επιτροπή αυτή ε, ε, συνεργαζόμενοι ε, λοιπώς. Οπότε δεν είναι πολύ ενθαρρυντική η κατάσταση, επιτρέψτε μου να συμπεράνω, αλλά μπορούμε να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε από την Επιτροπή μας να επιτύχουμε αποτελέσματα σημαντικά ώστε να καταγγείλουμε καθαρά, χωρίς περιστροφές, το πώς παραβιάζεται η συνεργασία από αυτούς τους μηχανισμούς, τις δομές που μπορεί μάλιστα να επιδεινώσουν τα προβλήματα που υπάρχουν, επηρεάζοντας σοβαρότατα την προστασία της, ε, των συμφερόντων του παιδιού. Εάν δεν δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα επιταχυνθούν οι δικαστικές αποφάσεις, απλά θα αποκρισταλωθεί μια κατάσταση ε, ε, όπως έχει αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη. Ε, για παράδειγμα, η Επιτροπή στις έξι αρχές που αναφέρει για την εκτελεστότητα του εξεκουάτουρ που θέλει να μελετήσει η Κομισιόνα διαγράφοντας τους ορισμένες περιπτώσεις θέλω να πω εξίσου σημαντική αν όχι περισσότερο είναι οι νέοι κανόνες για την προστασία και την ακρόαση του παιδιού αλλά και διατάξεις περί συνεργασίας μεταξύ κεντρικών αρχών σε θέματα γονικής ευθύνης. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη συγκέντρωση και την ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις που σχετίζονται με τους γονείς. Ε, κάτι σημαντικό για τη λήψη αποφάσεων ε, αναπερίπτωση και που έχουν σημαντικές επιπτώσεις ε, για το παιδί. Τέτοιοι κανόνες φαίνεται να καθοδηγούνται από θετικές προθέσεις αλλά αν τους επαληθεύσει κανείς ε, στις λεπτομέρειές τους ε, μπορεί να βρει ε, διακριτική μεταχείριση στους μηχανισμούς και στις πρακτικές οπότε αυτά πρέπει να ελεγχθούν σε επίπεδο κρατών μελών. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να οι παρεμβάσεις μας να καταλήξουν σε διέξοδο παρεμβάσεις οι οποίες φυσικά καθοδογούνται από ένα πνεύμα προστασίας των δικαιωμάτων ε, που προβλέπονται από τις διεθνείς συμφωνίες, από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καμία, κανένα περιορισμό των δικαιωμάτων αυτών. Είμαι βέβαιη ότι με τους συναδέλφους θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε και ευχαριστώ και τη συναδελφό Καμπεσάν που δεν είναι παρούσα για το πρώτο σχέδιο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Ντανούκα. Σας ευχαριστώ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις τροπολογίες του εισηγητή. Συμφωνούμε με κάποιες από αυτές. Ε, με τις 1, 2, 3, 4... Και αν κοιτάξουμε την τροπολογία 4, Αναφέρεται ότι χρειάζονται επαγγελματίες διαμεσολαβητές, ε, ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργοί. Δεν συμφωνώ απολύτως ε, με την τροπολογία 8, που είναι πιο συγκεκριμένη και μιλάει για το παιδί όταν είναι άνω των 13 ετών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η απόψει του παιδιού, ενώ άνω των 16 ετών οι επιθυμίε του θα πρέπει να θεωρούνται ω αποφασιστικέ. Έχω λοιπόν ερώτηση προ ε, την ε, αντικαταστάτρια του εισηγητή. Πώ καταλήξατε στις συγκεκριμένες ηλικίες όσον αφορά το να η υπόψη η, η γνώμη του παιδιού. Στην τροπολογία 5 αναφέρεται η οικονομική κατάσταση ενός γονέα και λέει ότι δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρείται ως καθοριστικό στοιχείο προκειμένου να εκτιμηθεί η ικανότητα του ή της να αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού. Όχι μόνο η οικονομική κατάσταση, αλλά και η υπηκότητα, η ηθαγένεια του γονέα. Πολύ συχνά ακούμε από αναφέροντες να δίδεται προτεραιότητα σε υπήκο του κράτους μέλους ε, όπου διαμένει το ζευγάρι. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να εισάγουμε και αυτό το στοιχείο στο κείμενο. Επίσης, αναφέρεται η γλώσσα. Αυτό είναι καλό. Διότι συχνά όταν ε, συχνά έχουμε αναφορές σε, σε περιπτώσεις ζευγαριών ε, ε, που μιλούν διαφορετική γλώσσα. Όσον αφορά την ε, παράγραφο 5 της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, συναντάμε τον άρθρο 64 παράγραφος 5 ε, αναφέρεται η έννοια της συνήθους διαμονής η οποία ορίζεται διαφορετικά στις διάφορες περιπτώσεις. Η έλλειψη λοιπόν σαφούς ορισμού του τόπου συνήθους διαμονής είναι πρόβλημα. Βλέπω ότι ο εισηγητής μας δεν είναι παρόν. Και τέλος, ε, συμφωνώ απολύτως ότι η θέση σε ισχύ της πρότασης θα πρέπει να είναι όχι 10 έτη μετά την ε, ημερομηνία εφαρμογής, αλλά την 5 ε, έτη μετά την ε, ημερομηνία εφαρμογής. Θα πρέπει ε, να εκπονείται η σχετική έκθεση. Να ευχαριστώ κυρία Στανόκα. Η κυρία Ροζιέρα απλά ε, αντικαθιστά τον ε, εισηγητή. Σας προτείνω να στείλετε κατευθείαν ένα mail κατευθείαν στον εισηγητή. Μα πώς να το εξηγήσω αυτό για τα 13 και 16 χρόνια. θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βίλαντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και κυρίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. που θίγει πάλι αυτό το θέμα. Και ευχαριστώ και για τις προτάσεις που έχουμε λάβει. Δεν μπορώ όμως να κρύψω, όπως και η κυρία Στανόκα, ότι αναρωτιέμαι σε τι βαθμό οι τροπολογίες σχετικά με το πεδίο, ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Ε, ήδη με την τροπολογία 5 έχω την εντύπωση ότι φεύγουμε από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Έχω αμφιβολίες για την τροπολογία 8, που επίσης ανέφερε η κυρία Στανόκα. διότι αναφέρονται οι ηλικίε των 13 και 16 ετών. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές νομικές παραδόσεις ε, στα κράτη-μέλη ε, σχετικά με την ηλικία από την οποία τα παιδιά μπορούν ε, να συνομιλήσουν με τον δικαστή, να ακουστεί η γνώμη τους. Το να θέλουμε λοιπόν συγκεκριμένα όρια ηλικίας παρεμβαίνει ε, στις εθνικές νομικές παραδόσεις. Και δεν έχουμε αρμοδιότητα να αλλάζουμε το ουσιαστικό δίκαιο στα κράτη-μέλη. Ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει τι είναι το καλύτερο για το παιδί. Και ουσιαστικά, όταν έχουμε διαζύγιο μεταξύ δύο Τσέχων, δύο Ιταλών, δύο Γερμανών, στο εθνικό δίκαιο. Εγώ γνωρίζω ε, από προσωπική μου πείρα ότι υπάρχουν ε, θέματα στα οποία οι νέοι βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά από ότι ένας αντικειμενικός τρίτος. Τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει τις ε, θέσεις τους στα στο δίκαιο της κάθε χώρας και δεν μπορούμε να επέμβουμε σε αυτό. Και τέλος, έχω αμφιβολίες και στο σημαντικό μεν θέμα της βίας με βάση το φύλλο, ε, το οποίο όμως δεν είμαι βέβαιος ότι έχει θέση εδώ. Ε, είναι σημαντικό το θέμα, αλλά ε, παρόλα αυτά ε, δεν μπορεί να παίρνει ξεχωριστή θέση ένα στοιχείο μόνο. Η εμπειρογνώμων, θα πρέπει να ε, ζητήσουμε την εμπειρογνωμοσύνη των ε, διαμεσολαβητών και των διαφόρων επιτροπών. Εδώ στην Επιτροπή Αναφορών έχουμε δει να ασχολούμαστε πολύ λίγο με το αν δικαστήριο τρίτης χώρας, παράδειγμα, ε, στο κράτος μέλος Α διαμένει η οικογένεια, στο κράτος μέλος Β λαμβάνεται απόφαση σχετικά με τη γονική μέρημνα και ε, ο γονέας με τη γονική μέρημνα πηγαίνει στο κράτος μέλος Γ και έτσι να αποκλείσει τον άλλον γονέα. Ο αποκλεισμένο γονέα προσφεύγει στο δικαστήριο και το δικαστήριο του κράτου μέλου Γ λέει δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι αποφασίστηκε στο κράτο μέλο Β. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των προβληματισμών μας. Ε, κάτι που ελάχιστα έχει γίνει στις τροπολογίες. Έτσι μπορούμε να κινήσουμε πολλά πράγματα, διότι ειδικά όσον αφορά την γονική μέρημνα όπου τα παιδιά ε, τραβιούνται στο δικαστήριο, δεν θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να ε, ε, ξαναανακρίνει τα παιδιά. Αυτές οι διαδικασίες επιβαρύνουν τα παιδιά και θα πρέπει στο βαθμό που είναι δυνατόν να περιορίσουμε αυτές τις διαδικασίες. Εάν δηλαδή έχει ε, εκδοθεί μια απόφαση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όλη την Ήπειρο. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ περισσότερο στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των ομιλητών ε, για το θέμα αυτό. Και η κυρία Ροσιέρ ε, μου είπε ότι ξέχασε να επισημάνει ότι πρόκειται για αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και οι τροπολογίες θα πρέπει να βασίζονται σε αναφορές που έχουμε λάβει για να μπορέσουμε να ε, συνεισφέρουμε στις εργασίες της επί της ουσίας αρμόδιας επιτροπής, της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων. Ε, και η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών είναι 9 ε, Μαρτίου στις 3 το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Πέτη θα γίνει 25 Απριλίου. Προχωράμε στο επόμενο θέμα γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 και φυσικά ο ρόλο τη Επιτροπή μα είναι ένα πολύτιμο κρίκο που συνδέει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με του πολίτε. Συναντάμε καθημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτε μα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Και χαίρομαι που μπορούμε να εκφράσω αυτό σε αυτή την γνωμοδότηση την οποία εκπονώ και φυσικά εξακολουθεί επί τη ουσία αρμόδια να είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Προετοιμάζει κάθε χρόνο μια έκθεση στην οποία καλούμαστε να συμβάλλουμε με τη δική μα γνωμοδότηση. Η προθεσμία για τροπολογίε είναι η 6η Μαρτίου η, στις 6 ε, το απόγευμα. στι 6 Μαρτίου. 6 το απόγευμα και η ψηφοφορία στη Γιούρη θα λάβει χώρα στις 12 Απριλίου. και στη δική μας επιτροπή στις 22 Μαρτίου. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες, ε, ε, διότι έχει περάσει η ώρα. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 10. Α, το 10 θα, το, θα περιμένουμε λίγο μέχρι να επιστρέψει ο επικεφαλής αντιπροσωπείας μας. Μπορούμε να περάσουμε στην αναφορά 1412 του 2015 σχετικά με το λογικοσμικό εξαπάτηση στα αυτοκίνητα. Ο αναφέρον δεν είναι εδώ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι η Μπάρμπαρα Μπονβισούτο. Και έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση σε σχέση με τις δράσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα Έχουμε εισαγεί ε, μια νέα διαδικασία έλεγχου ε, μέσω μιας δέσμης διαφορών νομοθετικών πράξεων, κανονιστικών πράξεων. Ο πρώτος και ο δεύτερος κανονισμός ε, για τις εκπομπές, τις πραγματικές εκπομπές, δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου και στις, του 2016 και στις 20 Απριλίου. Με τις δύο αυτές πράξεις η Κομισιόν έχει αναλάβει σημαντικά βήματα για τη μείωση του επίπεδου των ε, επιβλαβών εκπομπών για την ε, ατμόσφαιρα και με τη δεύτερη πράξη η Κομισιόν δεσμεύεται να ενεργοποιήσει την αναθεώρηση των ε, επωνομαζόμενων συντελεστών συμμόρφωσης που αναφέρονται στην αναφορά ετησίως ώστε αυτοί οι συντελεστές συμμόρφωσης, ο συντελεστής συμμόρφωσης να, έρθει, να φτάσει στο ένα το σύντομότερο δυνατόν. Η Κομισιόν έχει προτείνει και μια τρίτη πράξη που επίσης θα μειώσει τη διαφορά μεταξύ των αριθμών μικροσωματιδίων που μετρώνται στο εργαστήριο και στο δρόμο. Η πράξη αυτή ψηφίστηκε από την Τεχνική Επιτροπή που αποτελείται από τα κράτη-μέλη το Δεκέμβριο πέρυσι και αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό εξέταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και τώρα μελετάμε την τέταρτη κανονιστική πράξη που θα ενισχύσει την επιτήρηση της αγοράς και που θα συμπεριλαμβάνει το δοκιμέ από ανεξάρτητα εργαστήρια τον περασμένο Ιανουάριο. Επίσης η Κομισιόν υιοθέτησε κατευθύνες γραμμές για την αξιολόγηση των στρατηγικών μείωσης των εκπομπών των αυτοκινητοβιομηχανιών περιλαμβάνουν και μεθόδους που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να εντοπίζουν πιθανές ε, ε, ύποπτες περιπτώσεις. Τέλος, η Κομισιόν συλλέγει στοιχεία για να αξιολογήσει την πρόοδο στα ΠΑΜΣ, τα φορητά συστήματα μέτρησης εκπομπών. Εκεί, όπως ανέφερα, υπάρχει ήδη μια ρήτρα αναθεώρησης στο δευτερεύουσα πράξη, οπότε βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνουμε, θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε μια αναθεώρηση των συντελεστών συμμόρφωση ε, όπως διατυπώνονται στη δεύτερη πράξη. Ε, αυτά από πλευρά μου. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε το λόγο στου συναδέλφους. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή απαρίθμησε όλα τα όμορφα πράγματα που φαίνεται να έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια Σήμερα, σήμερα, ακριβώ πριν μια ώρα ψηφίστηκε η τελική έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής ΕΜΙΣ που δημιούργησε το Κοινοβούλιο φέτος για την έρευνα του σκανδάλου. Μάλιστα, ένα στοιχείο, οι συντελεστέ συμμόρφωση εισήχθησαν ουσιαστικά για να διπλασιαστούν τα όρια εκπομπών οξυδίων του αζότου χωρί καμία επιστημονική βάση. Αναγνωρίζεται εκ των πραγμάτων και στην τελική έκθεση ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν επιμείνει, όπως έχουν επιμείνει και πολλά κράτη-μέλη και το δικό μου και η Ιταλία, στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής όπου ουσιαστικά βοηθάμε να χαθεί χρόνος μέσω της εισαγωγής αυτών των τεστ, των RD, εισάγοντα συντελεστέ συμμόρφωση, πολλαπλασιαστέ, υπερβολικά υψηλού, πολύ ψηλότερου σε σχέση με αυτό που αντικειμενικά είναι απαραίτητο. Ξέρετε και στη διάρκεια των ακροάσεων που οργανώσαμε στην Επιτροπή, εμείς όλοι οι τεχνικοί προγνωμόνες επιβεβαίωσαν ότι τα όρια ήδη σήμερα είναι δυνατόν να τηρηθούν σε πραγματικές συνθήκες. Η Αμερικανική νομοθεσία, για παράδειγμα, είναι πολύ πιο αυστηρή από την Ευρωπαϊκή και παρόλα αυτά τηρείται. Οπότε από τεχνική άποψη δεν υπάρχει απολύτως καμία ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πολλαπλασιαστές συμμόρφωσης. Εγώ συμφωνώ με τις ανησυχίες των αναφερόντων σε αυτές τις αναφορές. Εύχομαι η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Διότι παρότι ψηφίστη, είχαμε την ψηφοφορία σήμερα, που έχουμε πολύ από το να καταλήξουμε σε μια επίλυση της κατάστασης. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα θεωρητικά, αλλά στο δρόμο στις πόλεις μας, στους δρόμους μας, θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν για δεκαετίες αυτοκίνητα, τα οποία συνεχίζουν να ρηπαίνουν ε, έως και κατά 90% περισσότερο από ό,τι επιτρέπεται. Η κατάσταση δηλαδή είναι δραματική. Επηρεάζει σημαντικότατα την υγεία των πολιτών, διότι μην ξεχνάμε στην Ευρώπη ετησίως ο αρμόδιος οργανισμός μας λέει ότι πρόωρα πεθαίνουν 450.000 άτομα. Είναι τρομακτικά τα νούμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την κατάσταση, να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε ποιος έχει τις ευθύνες, διότι σήμερα κανένας δεν ε, πληρώνει το τίμημα. Ε, σε κανέναν δεν ε, ε, επιβάλλονται κυρώσεις ε, για να εισακουστούν οι πολίτες. Ε, ούτε αποζημιώσεις προς τους πολίτες έχουμε όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε έχουμε δύο κατηγορίες πολιτών στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε ενώπιον ενός προβλήματος στο οποίο, στο οποίο κάνουμε τα στραβά μάτια. Ελπίζω οι αναφορές να παραμείνουν ανοιχτές και πιστεύω ότι πρέπει να σταλούν και προς ενημέρωση στις Επιτροπές Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Μεταφορών, Επιτροπές που είναι αρμόδιες επί του θέματος σήμερα. Ευχαριστώ, Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ πολύ. Με λίγο πικρόχολο χιούμορ. Θα μπορούσα να πω ότι είναι θλιβερό το ότι συχνά χρειαζόμαστε πρώτα την καταστροφή για να διορθώσουμε την κατάσταση. Και επίση ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να βελτιώσουμε τη στατιστική ή την πραγματικότητα. Ε, αλλά ε, συχνά κρύβονται τα στοιχεία στην στατιστική και χάνουμε από τα μάτια μας την πραγματικότητα. Και η καινοτομία στο λογισμικό προφανώς έχει ε, πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο και όχι στην πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν ε, καλά και κακά νέα. Χαίρομαι που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει την πραγματικότητα. Δεν είναι ε, απλή η κατάσταση και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά να σταλεί στην ε, αρμόδια επιτροπή. Ε, και δεν θα πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας. Χρειαζόμαστε σωστές τιμές στην πραγματικότητα, ρεαλιστικές τιμές όμως. Και από τις υποθέσεις των προηγουμένων ετών θα πρέπει να μάθουμε, να αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και να την στείλουμε στην αρμόδια επιτροπή. Εάν ε, δεν ε, γίνει τίποτα, αν δεν ακούσουμε τίποτα μπορούμε να την κλείσουμε, αλλά σήμερα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. You can give the floor to Mrs. because she asked it uh, at the beginning and then me. Δώστε το λόγο στην κυρία Άουκεν γιατί τον είχε ζητήσει προηγουμένως, νωρίτερα από μένα. Μάργαρετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Νότι. Θα ήθελα να πω ότι είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ο Πίτερ ζήτησε να παραμείνει αναφορά ανοιχτή. Να το σημειώσουμε στα πρακτικά. Παρακαλώ. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω μείνει άφωνη. Έχω μείνει άναυδη. Ζητήσατε να μείνει ανοιχτή. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή και πρέπει να το πούμε είναι μία από τις πιο βλαπτικές υποθέσεις στη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αίσθηση, αυτή η φήμη ότι δεν ακολουθούμε τη δίκαιη μεταχείριση, τις προσταγές της επιστήμης, δεν τηρούμε και δεν μεριμνούμε για την ασφάλεια των ανθρώπων, δεν τηρούμε καν τους, κανού, τους καλούς κανόνες για το διεθνή ανταγωνισμό. Υπονομεύουμε τη δυνατότητα που έχει η βιομηχανία μας η ευρωπαϊκή να γίνει ταγό σε διεθνές επίπεδο και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο και όλο το ευρωπαϊκό σύστημα θα ανταποκριθούν με έναν τρόπο ο οποίος ίσως μπορέσει να ξανααποκτήσει, ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη ε, στον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος. Και γι' αυτό στηρίζω τον Πίτερ. Συμφωνώ δηλαδή με αυτά που είπε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν ξέρω ε, ποια είναι η έκβαση στην Επιτροπή εμείς σήμερα. Ωστόσο, να ασκήσουμε πίεση. Ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η χειρότερη. Η κακή ήταν και η πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Αλλά αν μπορούμε να προχωρήσουμε αυτό θα είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά. Ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο βεβαίως απασχολεί την Ευρώπη, απασχολεί πάρα πολλές χώρες και νομίζω ότι αναδεικνύει τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν κατά το παρελθόν. Ο τρόπος ελέγχου όλου του συστήματος αυτού διότι αποδείχθηκε ότι ο έλεγχος δεν ήταν αποτελεσματικός, αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αποδείχθηκε ότι δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη αυτοκινητοβιομηχανία, ε, αλλά και άλλες, διότι το ζήτημα είναι ανοιχτό. Είχα υποβάλει και σχετική ερώτηση ε, στην ε, Κομισιόν και από την απάντηση προέκυπτε ότι δεν αφορά μόνο ότι ε, υπόθεση Volkswagen, αφορά και άλλες υποθέσεις άλλων ε, εταιριών ευρωπαϊκών Επομένως νομίζω ότι είναι σοβαρό το ζήτημα. Έχουμε βέβαια ως Κοινοβούλιο μια ειδική επιτροπή η οποία ασχολείται με το θέμα αυτό. Προφανώς έχει αυξημένες αρμοδιότητες και αυτή έχει και την, ε, αν θέλετε, την τεχνογνωσία πλέον με τους ε, ε, εξπέρ που έχει κοντά της, τους πραγματογνώμονες, τον τρόπο με τον οποίο θα εξετάσει. Δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, δεν γνωρίζω την εξέλιξη, αλλά σίγουρα εμείς ως Επιτροπή, οφείλουμε να, Επιτροπή Αναφορών, οφείλουμε να κρατήσουμε ανοιχτή την υπόθεση, οφείλουμε να πιέσουμε παραπέρα την ίδια την Κομισιόν για πολύ πιο σοβαρές μελέτες και παρεμβάσει, να πιέσουμε αν θέλετε και την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου που εξετάζει αυτά και να δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται διαφάνεια και πρέπει να στηρίξει τα αιτήματα των πολιτών, πρέπει να στηρίξει τα θέματα ε, της προστασίας του περιβάλλοντος, πρέπει να στηρίξει την, ε, τα ζητήματα που αφορούν την υγεία των ίδιων των πολιτών. Επομένως νομίζω ότι έχουμε πλήρη συμφωνία να παραμείνει παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να αναμείνουμε τις εξελίξεις και εν συνεχεία να ξαναέρθει η υπόθεση σε εμά για να δούμε πώς μπορούμε να τη χειριστούμε ακόμη πιο καλά. Ευχαριστώ. Thank you very much. And I also agree. I think that this is the way to, to move forward. We need to... Πράγματι, συμφωνώ και εγώ. Αυτός είναι ο τρόπος να προχωρήσουμε, να δούμε ε, πώς θα προχωρήσει το θέμα στην Επιτροπή. Εμείς, στην Ειδική Επιτροπή, που το συζητά, διατηρούμε λοιπόν την αναφορά ανοιχτή και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περισσότερα στοιχεία μετά από την ψηφοφορία στην ΕΜΙΣ. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε και με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που, με τους οποίους οι απόψεις μας συμπίπτουν από καιρού εις καιρών. Και αυτό μας ενθαρρύνει και μας αναζωογονεί, ότι με όλους μπορούμε να έχουμε απόψεις που να ε, συμπίπτουν και μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους λοιπούς και την Ελεονόρα βεβαίως. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Ζητώ συγγνώμη γιατί Κινήθηκα πολύ γρήγορα όσον αφορά τη δική μου γνωμοδότηση για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το 2015. Είδα ότι κάποιοι είχαν αποχωρήσει από την αίθουσα. Νομίζω ότι για τις νομοδοτήσεις δεν πρέπει να περνάμε υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην καθυστερούμε, εκτός και αν είναι κάτι το πραγματικά κρίσιμο. Έχουμε αναφέροντες που περιμένουν. Να προχωρήσουμε στο επόμενο ζήτημα. Η επόμενη αναφορά είναι η 987 του 2015 για την αλλαγή στους ε, καταλήτες και το σχετικά συστήματα επιλογής και διαλογής μετά την υπόθεση την, της Volkswagen. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυρία Μπονβισότο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, βεβαίω η αναφορά αυτή σχετίζεται άμεσα και με την προηγούμενη. Να προσθέσω λοιπόν ότι Αυτές οι συσκευές απαγορεύονται από το 1998 και οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν την υποχρέωση βεβαίως να τηρούν το νόμο και σύμφωνα με το σημερινό σύστημα εγκρίσεων τύπου αρμοδιότητα για την απαγόρευση έχουν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη το είπα, έχει προτείνει ε, μια νέα διαδικασία δοκιμής και δοκιμασίας των εκπομπών. Το είχε προτείνει πριν αποκαλυφθούν και οι χειραγωγήσεις ε, των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Ε, έχω επενθυμίσει ήδη την πρόταση του Μαΐου του 2015, μετά επιταχύναμε τις προσπάθειές μας για να ολοκληρώσουμε το πακέτο προτάσεων. Είχαμε την έγκριση του RD2, εξετάζεται το RD3 και θα ακολουθήσει και το RD4. Με τη θέσπιση αυτών των δοκιμών στους δρόμους, ο κίνδυνος εξαπάτησης με συσκευές τέτοιου τύπου θα ελαχιστοποιηθεί. Βέβαια δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται επαρκής και αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016 ε, πρότεινε ένα ε, συνολικό σύστημα εγκρίσεων τύπου για να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα και ανεξαρτησία μεταξύ των διαφόρων συστημάτων δοκιμών, να υπάρχει μεγαλύτερη επιτήρηση εποπτεία οχημάτων και μεγαλύτερη αναγνώριση του ρόλου της. Θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή θα καλύψει τις αδυναμίες του φυστάμενου συστήματος και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν την πρότασή μας το συντομότερο δυνατόν και να αρθούν στο δικό μας επίπεδο φιλοδοξίας το οποίο είναι υψηλό. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση έναντι 7 κρατών μελών γιατί δεν εκπλήρωσαν τις προ υποχρεώσεις τους ε, σε σχέση με τις εκπομπές ε, των αυτοκινήτων και τις ε, ταξινομήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε το λόγο των συναδέλφους. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Ελεονόρα, ναι, ήθελα να προσθέσω απλά. Πράγματι, οι συσκευές εξαπάτησης απαγορεύονται. Ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις όσον αφορά τη χρήση ε, συσκευών ελέγχου των ε, εκπομπών στα οχήματα και εκεί είναι το πρόβλημα διότι οι επιχειρήσεις, οι κατασκευαστές μεταξύ των οποίων η Volkswagen αλλά και άλλοι επικαλούνται αυτές τις εξαιρέσεις που ουσιαστικά μειώνουν ε, την αποτελεσματικότητα των λογισμικών ε, που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση αυτών των εκπομπών, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να υποστεί ε, βλάβη ο κινητήρας. Σε μια ακρόαση μας έλεγε κάποιος ότι για να αποφευχθεί πιθανή διακοπή της λειτουργίας του οχήματο κατά την οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ε, διαφορετικά αυτές οι στρατηγικές ε, καταπολέμησης των εκπομπών. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Volkswagen ε, παραδέχτηκε την εξαπάτηση. Στην Ευρώπη κανεί δεν το παραδέχεται, αλλά συντρέχουν όλες οι προποθέσει για να συνεχιστεί η έρευνα και για να αντιληφθούμε επιτέλους ότι έπαιξαν όχι μόνο με την εμπιστοσύνη των πολιτών αλλά και με την υγεία τους. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Οπότε λέω να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά όπως και την προηγούμενη και να ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία όπως με την προηγούμενη αναφορά. Πέτερ Ο Πέτερ Όχι, ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Μαριάς ζήτησε το λόγο πρώτος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ε, η αναφορά αυτή έχει άμεση σχέση και με όσα υπόθηκαν και από τη δική μας πλευρά για την προηγούμενη αναφορά ε, θέλω σε αυτό το σημείο να επιμείνω στην πλευρά της εξαπάτησης των καταναλωτών, διότι έχουμε την Volkswagen η οποία παραδέχθηκε πράγματι όσον αφορά τις ΗΠΑ ότι εκεί υπήρξε μια εξαπάτηση των καταναλωτών και ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία για την αποζημίωσή τους. Το ίδιο βεβαίως πρέπει να γίνει αποδεκτό και στην Ευρώπη, διότι έγινε εξαπάτηση των καταναλωτών και στην Ευρώπη από την Volkswagen με την παραποίηση των στοιχείων, με όλη τη διαδικασία αυτή, με το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, αυτή τη στιγμή που υπάρχει ομολογία της εταιρεία ότι εξαπάτησε τους καταναλωτές της ΗΠΑ, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συζητούμε επιδερμικά το ζήτημα αυτό και πρέπει να συζητήσουμε την ουσία. Πώς δηλαδή οι ίδιοι οι καταναλωτές θα αποζημιωθούν από την ε, Volkswagen για την εξαπάτηση την οποία επέστησαν Και ταυτόχρονα να δούμε και τις επιπτώσεις στην υγεία των ίδιων των καταναλωτών αλλά και στη δημόσια υγεία. Επομένως οφείλει η Κομισιόν να συνεχίσει πολύ πιο αποφασιστικά τη δραστηριότητά της αλλά και τα κράτη-μέλη, γιατί και αυτά έχουν ευθύνη, να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα, ούτω ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική τιμωρία. Να μην ξαναγίνει αυτό από την πλευρά τη Volkswagen. Όμω, επιμένω ότι είναι θέμα να εξεταστούν και οι άλλε ευρωπαϊκέ αυτοκινητοβιομηχανίε, διότι στην απάντηση που σας είπα, που έλαβα σε ερώτηση που έκανα προς την Κομισιόν για την υπόθεση Volkswagen, απαντήθηκε ότι και άλλες εταιρείες ευρωπαϊκές ε, επίσης εξετάζονται και ελέγχονται για το κατά πόσο και αυτές εξαπάτησαν τους ίδιους τους καταναλώτες. Άρα λοιπόν είναι ένα σοβαρό θέμα να μείνει ανοιχτό και να, έχουμε την, να στηρίξουμε πλήρως τους αναφέροντες σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Now... Ευχαριστούμε πολύ. Πέτρα, έχετε το λόγο. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά να την στείλουμε και στην ε, Ειδική Διερευνητική Επιτροπή. Και περιμένω και συστάσεις από την ε, Επιτροπή αυτή σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, προστασία των καταναλωτών. καλά το είπα, αλλά όσον αφορά την αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις, οι Αμερικανοί μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Θα πρέπει σε περίπτωση που ε, ανακαλύπτεται μια απάτη να υποβάλλεται ε, αποζημίωση. Δηλαδή, εάν ε, εξαπατώ κάποιον, θα πρέπει να γνωρίζω ότι αν με πάρουν χαμπάρι θα πονέσει η τιμωρία. ελπίζουμε λοιπόν ότι από την Διαρνητική Επιτροπή θα έχουμε και βελτίωση της νομοθεσίας. Και θα μπορέσουμε να κλείσουμε την αναφορά όταν κλείσει και η, αναφορά, η Επιτροπή της ε, Εργασίας της. Ε, πάντως ε, από την κρίση αυτή έχουν δημιουργεί και κάποιες ευκαιρίες. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω ότι η Επιτροπή εμείς ε, κλείνει αυτή τη στιγμή, διότι μετά την ψηφοφορία κλείνει και η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της. Ε, αλλά ας κάνουμε το εξής, ας αφήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και να παραμείνουμε σε διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και θα παρακολουθήσουμε και τις διαδικασίες περιβάση στα τα κράτη-μέλη που αναφέρατε αρχικά. Ε, ωραία, αυτό ας κάνουμε και να προχωρήσουμε. Είναι χαρά μου και τιμή μου να καλωσορίσω τους αναφέροντες ε, για την ε, αναφορά 1328 κάθετος 2015 ε, του Ρενάτο Αμορότο σχετικά με το καθεστώς των ειρηνοδικών στην Ιταλία και μια άλλη σειρά αναφερόντων καλωσορίζω. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στους αναφέροντες σε πέντε λεπτά τον καθένα ξεκινώντας από τον Ρωσέλα Μπαρόνε. Αξιότιμη πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, το άτομα για άνοιγμα διαδικασία επί παραβάση εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντί τη Ιταλία για την παράνομη μεταχείριση των επίτιμων δικαστών και ειδικότερα των ειρηνοδικών βασίζεται στην επαναλαμβανόμενη κατάχρηση των συμβάσεων την τελευταία 20 ετία όπως εφαρμόζονται για την κατηγορία επαγγελματιών τη δική μα που έρχεται σε αντίθεση με ε, τις διατάξεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η θέση των ειρηνοδικών έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 70 του 99, μέσα στην οποία το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει τη Συμφωνία Πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου. Η Συμφωνία Πλαίσιο, όπως προβλέπεται, καθορίζει τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες απαιτήσει που σχετίζονται με την εργασία ορισμένου χρόνου. Επίσης αναφέρει τη βούληση των κοινωνικών ε, εταίρων να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο που καθορίζει την εργασία των εργαζομένων ορισμένου χρόνου προστατεύοντάς τους από τη διακριτική μεταχείριση. Η Ιταλική νομοθεσία σε σχέση με τους ειρηνοδίκες παραβιάζει το πλαίσιο αυτό σε τρεις περιπτώσεις αιτιολογεί αδικαιολόγητα ε, μια εργασιακή σχέση λανθασμένη και υπέρβαση των ορίων διάρκειας ανανέωσης των, ε, ε, της απασχόλησης. Η αιτιολόγηση της αυτής εργασιακής σχέσης υποτίθεται ότι οδηγεί στην κάλυψη προσωρινών αναγκών. Οι συμβάσει αυτέ ορισμένου όργου ε, έργου τελικά καλύπτουν μόνιμες απαιτήσει των εργοδοτών και πρέπει να θεωρηθούν καταχρηστικές. Να υπενθυμίσουμε την απόφαση C21204 της 4 Ιουλίου του 2006 για τις καταχρήσεις εδώ και 15-20 χρόνια από το δικαστικό σύστημα πολλών επίτιμων δικαστών και ερηνοδικών. Ε, σε αστικές υποθέσεις και σε ποινικέ υποθέσεις. Ε, η Ιταλική νομοθεσία έρχεται σε αντίθεση και με τη Συμφωνία Πλαίσιο όπου δεν ε, υπάρχουν λόγοι που να αιτιολογούν την ανανέωση των συμβάσεων. Η, η απόφαση του 2010 λέει ότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να είναι γραπτή και να αιτιολογεί την ύπαρξη της σύμβασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται θα πρέπει να μην ισχύει η ημερομηνία ε, λήξης ισχύω της σύμβασης. Σε καμία περίπτωση η Ιταλική κυβέρνηση δεν έχει αιτιολογήσει την επανάληψη, την ανανέωση αυτών των συμβάσεων. Συμπερασματικά η Ιταλική κυβέρνηση ενώπιον ημών των επίτιμων δικαστών και ειρηνοδικών παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο με την καταχρηστική ανανέωση των συμβάσεων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση και να ζητηθεί από το Ιταλικό κράτος να προβλέψει τη σταθεροποίηση, τη μονιμοποίηση αυτής της κατηγορίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο με ίση αμοιβή όπως αυτή των έμειστων δικαστών με τις κλασικές εγγύησεις για τους εργαζομένους του δημοσίου τομέα, με την ε, κάλυψη ε, ασθενείας ε, και συνταξιδοτική κάλυψη και της άδειας Εγώ ως μητέρα δύο δίδυμων ε, και πολλές συναδελφοί μου αποτελέσαμε το αντικείμενο εκμετάλλευσης καθώς χρειάστηκε να ε, ξαναπιάσουμε δουλειά δύο μήνε μετά τη γέννηση. Για να μην μιλήσω για του αδέρφου που κατά διάρκεια χημειοθεραπεία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη δουλειά του. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο δίνουμε τώρα στην Μανουέλα Αρτόνα, επίσης για πέντε λεπτά. Καλημέρα. Ονομαζόμαι Εμμανουέλα Αρτόνα, ειρηνοδίκη στη Ρώμη επίτιμος ονομάζομαι από το 1998. Από 19 χρόνια, δηλαδή με ειρηνοδίκη 15 χρόνια, χωρίς διακοπή και με σε πλήρη αποσχόληση. Ασχολούμαι με 5.000 υποθέσεις ετησίως και αυτό δεν μου επιτρέπει να διεξάγω καμία άλλη εργασία. Ω ειρηνοδίκης έχω διεκπαιρεώσει πάνω από 10.000 υποθέσεις αστικές και ποινικές. Είναι πλασματική, πλασματικός ο χαρακτηρισμός επίτιμος για τους ε, ειρηνοδίκες που υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα επίτιμο. Ο ίδιος ο Ιταλός νομοθέτης αυτό διαψεύδεται στο άρθρο 11.4 του νόμου 374 του 91 υπάρχει ε, ανώτατο όριο αποφάσεων που ανταμείβονται από το κράτος για τον Ειρηνοδίκη στις 2000 και κάτι ε, που είναι ο ίδιος αριθμός που απαιτείται από έναν έμιστο δικαστή. 56 περίπου ευρώ είναι η ανταμοιβή, η μετριόπατη ανταμοιβή προς, τους, προς εμάς. Και ξέρετε, οι αποφάσεις των ειρηνοδικών έχουν την ίδια αξία με ε, αυτές των τακτικών δικαστηρίων. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο ότι αντικειμενικά για να διεκπαιρώσει κανείς 1267 ε, αποφάσει πρέπει να δουλεύει σε πλήρες ε, ωράριο και δεν έχει χρόνο για καμία άλλη απασχόληση. Πρέπει να είναι επαγγελματίας, ο ειρηνοδίκης, παγιωμένος μέσα στο χρόνο, και δεν είναι τυχαίο που ανανεώνονται οι θητείες μέχρι και 20, σε 20 χρόνια. μετά από έγκριση της καταλληλότητας τους από τα διάφορα αρμόδια συμβούλια. Το Ιταλικό κράτος έχει ορίσει λοιπόν τον όρο στις 1267 αποφάσεις το χρόνο η παραγωγή των επίτιμων δικαστών ουσιαστικά, ε, καθώς εργάζονται με πλήρες ωράριο, είναι πολύ υψηλή, ε, με κόστος γελίο για το Ιταλικό κράτος, καθώς ε, στερούνται οποιασδήποτε προστασίας στο πλαίσιο εμείς της εργασίας. Το Ιταλικό κράτος ανανεώνει διαρκώς τις θητείες των λόγω επίτιμων δικαστών για 10-20 χρόνια χωρίς διακοπή ώστε να μην παραλύσει το Ιταλικό δικαστικό σύστημα που σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές ε, απασχολεί για το 50% των υποθέσεων αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν κανένα εργασιακό προνόμιο. Βάσει διαφόρων αποφάσεων έχει αναγνωριστεί ήδη ε, συμπερασματικά ο νόμος 374 του 91 και οι παρατάσεις ε, των ε, θητιών και αυτός ο τίτλος του επίτιμου δικαστή έχει επιτρέψει την εκμετάλλευση των εργαζομένων αυτών από το Ιταλικό κράτος με γελίο κόστος καθώς ε, δεν έχουν καμία προστασία, κανένα δικαίωμα, ε, όπως συμβαίνει με την έμειστη συνεργασία. Με την αναφορά αυτή ζητάμε να επιβεβαιωθούν αυτές οι παραβιάσει του Ιταλικού κράτους, να ξεκινήσει η διαδικασία επί που προβλέπονται από τα άρθρα 258 και 260 της συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε και τώρα καλό θα ήταν να ακούσουμε και την Ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία Νίκολα Μινάση είναι ο συντονιστή για τι διαδικασίε παραβάση και την κρατική βοήθεια και να σα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίξτρομ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, αξιόμενοι αναφέροντες, ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η υπόθεση. Έχει διαρκέσει πολύ καιρό και έχει την την προσοχή της Ιταλικής κυβέρνησης. Η υπόθεση για την οποία συζητάμε και που έχει δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες ε, βασίζεται στο ότι έγιναν προσπάθειες ε, να βρεθεί ένας τρόπος ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επίτιμων δικαστών και των έμιστων δικαστών. Αυτό κατέστη αδύνατον στην πραγματικότητα καταρχάς για ένα νομικό λόγο το Ιταλικό Σύνταγμα ε, θεσπίζει ότι η δικαστική λειτουργία ασκείται από έμεστους δικαστές και το, ο θεσμός του επίτιμου δικαστή προβλέπεται επικουρικά από προσωπικό ε, πιστοποιημένο για την εργασία σε δικαστήρια και χαρακτηρίζεται ε, επικουρική εργασία που δεν μπορεί να οδηγήσει σε ε, δικαστική εξίσωση ε, με την ε, λειτουργία του ΕΜΙΣ δικαστή. Οι εμείς οι δικαστές μάλιστα ε, επιλέγονται με διαγωνισμό ενώ οι επίτιμοι με συνέντευξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επίτιμοι δικαστές δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Φυσικά και διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για τη λειτουργία των Ιταλικών δικαστηρίων και γι' αυτό το λόγο η Ιταλική κυβέρνηση θέλει οπωσδήποτε να αναγνωρίσει ε, σε αυτούς η συμμεταχείριση με αυτή των έμιστων δικαστών. Όσον αφορά την αμοιβή, το δικαίωμα ίδιας μητρότητας, ε, το δικαίωμα ε, για διακοπές, ε, για άδεια διακοπών και αποδεκτά ωραία εργασίας. Συμφέρει την Ιταλική κυβέρνηση να βρει μια λύση η οποία θα επιτρέψει την αναγνώριση της ίσης μεταχείρισης και φυσικά αυτό θα πρέπει να βρει σύμφωνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει ξεκινήσει λοιπόν ένας διάλογος όπου η Ιταλία θα εξετάσει να δει πώς μπορεί να βρει αυτή την ισορροπία και να προβεί σε ταχύ επανακαθορισμό της κατάσταση του τομέα αυτού, ώστε να επιληθούν τα προβλήματα. Και αυτό μάλιστα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπήγοντο, διότι η κυβέρνηση έχει νομοθετική εντολή από το Κοινοβούλιο της Ιταλίας, η οποία θα εκπνεύσει το Μάιο. Οπότε η Ιταλική κυβέρνηση έχει κάθε συμφέρον να βρει γρήγορα μια λύση που να επιλύει και τα αιτήματα αυτά τα οποία μόλις ακούσαμε. Εμείς βλέπουμε λοιπόν πολύ θετικά την ε, ε, συζήτηση με την Κομισιόν, γίνονται επαφές και από πλευράς κυβέρνησης προτιθέμεθα να βρούμε μια ικανοποιητική λύση. Γρήγορα, μέχρι το προθεσμία του Μαΐου. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστούμε πολύ. Η Κομισιόν βρίσκεται εδώ. Η Ντάνα Τραμαζάντα παρακολουθεί έχει το λόγο να μας εξηγήσει την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά βεβαίως την κατάσταση που περιγράψατε Έχουμε ήδη δεχθεί πάρα πολλά παράπονα, περίπου 70 προσφυγές έχουμε δεχθεί. Ε, Πολύ σοβαρή υπόθεση φαίνεται. Πάρα πολλές λεπτομερείς πληροφορίες έχουμε λάβει, εκατοντάδες σελίδε που συνεχίζουμε να αναλύουμε και να εξετάζουμε. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ιταλικής Αντιπροσωπείας, συνεργαζόμαστε στενά με τις Ιταλικές Αρχές για την εξέβρεση λύσης. Σε αυτό το στάδιο το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συνεχίζουμε να αναλύουμε την Ιταλική νομοθεσία τις προσφυγές, τα, τις πληροφορίες που έχουμε λάβει. Να πω ότι θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα εξής ζητήματα στον ορισμό στο, του εργαζομένου, το δικαίωμα στην άδεια μητρότητα, στο, τη καταχρηστική προσφυγή ε, στα συμβάσει ορισμένου χρόνου και η μη διάκριση μεταξύ των συμβασιόχων του χρόνου και ορισμένου χρόνου μεταξύ άλλων. Και ελπίζουμε με όλα αυτά να γρήγορα να έρθουμε σε μια καλή λύση για τους ε, επιτιμή δικαστές. Είναι περίπου το 40% των ε, υποθέσεων που εντάσσονται στο Ναστικό κώδικα, δεν είναι μικρή δουλειά. Ελπίζουμε να φτάσουμε σε μια γρήγορη λύση και ικανοποιητική. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ γιατί είστε ακριβείς και ε, δεν ξεπεράσατε το χρόνο και μιλήσατε με νούμερα και στοιχεία και με ακρίβεια. Ο κύριος Κοζολίνο ασχολείται ιδιαίτερος με το ζήτημα αυτό και το ερώτημά σας έχει, μας έχει διαφωτίσει. Θα πάρετε εσείς πρώτα το λόγο. Παρακαλώ. Προσωπικά υποστηρίζω τη θέση που παρουσίασαν εδώ οι αναφέροντες και εγώ έχω απευθύνει ερώτημα προς την Κομισιόν ε, και η απάντηση που λαμβάνω εν μέρη απόψε ε, αντιστοιχεί στις κατευθύνσεις που έχω αποφασίσει και εγώ για το θέμα αυτό. Τώρα, επειδή εδώ δεν ήρθαμε να συζητήσουμε επί της ουσίας να βρούμε λύσεις, ε, δεν είναι δικός, δική μας αρμοδιότητα, εμείς μπορούμε να κάνουμε όμως το εξής. Αυτή είναι η δική μου έκκληση προς εσάς, προς όλους τους συναδέλφους Ιταλούς και εμεί να προωθήσουμε μια πρωτοβουλία μέσω μιας επιστολής στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στην αντίστοιχη Επιτροπή και στην Επιτροπή ώστε φυσικά να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά αυτό είναι αυτονόητο, δεν μπορούμε να την κλείσουμε αλλά να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το παραθράκι που έχει ανοίξει. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει προθεσμία μέχρι το Μάιο. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να δώσει μία απάντηση επί της ουσίας και πιστεύω ότι ε, έτσι πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διατηρήσει ανοιχτή την ε, αναφορά και να ζητήσει από τα ε, μέρη τον Αρμοδιοπουργό, την Επιτροπή και με την πλήρη συμμετοχή των αναφερόντων, διότι στην Ιταλία όταν συναντήθηκαν ε, στις σχετικές συνεδρίες δεν είχαν κληθεί, δηλαδή να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι και οι εκπρόσωποι ώστε να βρεθεί μια λύση. Είναι εμφανές ότι μετά από τόσα χρόνια που έχουμε στην πλάτη μας, ξεκινώντας από το 91, μιλάμε για 15-20 χρόνια, παραπάνω μάλιστα, είναι προφανές ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αν μη τι άλλο, διότι αυτή επιτελούν ε, έναν σημαντικότατο ρόλο στη δεκπεραίωση του τεράστιου όγκου υποθέσεων που έχει να αντιμετωπίσει η αστική δικαιοσύνη στην Ιταλία. Οπότε ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. ο κίνδυνος του να υπάρχει μια διαρκής διένεξη μεταξύ του κοινοτικού δικαίου, του εργατικού δικαίου, του Ιταλικού συντάγματος και των διαδικασιών επιλογής προσωπικού για το θέμα αυτό υπάρχουν επαρκείς αιτίε για να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιήσει τους ειρηνοδίκης στην Ιταλία που απαιτούν δικαίως ε, τα δικαιώματά τους και έτσι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε και ένα αρχαιότατο πρόβλημα που έχουμε στην Ιταλία τις καθυστερήσεις ε, ε, στη διεκπαιρέωση των υποθέσεων, ειδικότερα στον αστικό τομέα. Οπότε εγώ θα έλεγα να κάνουμε μία επιστολή ως Επιτροπή Αναφορών βάσει των όσων ακούσαμε και των αναφορών που έχουμε λάβει από του αναφέροντε και να ζητήσουμε από την Κομισιόν και από την Ιταλική κυβέρνηση μέσα στι επόμενε εβδομάδε να καταβάλουν κάποιε προσπάθειε ώστε να καταλήξουμε σε μια πρόταση μέχρι τα τέλη του Μαΐου και μετά να καλέσουμε ξανά ε, την Επιτροπή Αναφορών να συζητήσει αυτό το θέμα, να ακούσει του πρωταγωνιστές και να δει κατά πόσο η λύση στην οποία έχουμε καταλήξει ικανοποιεί του αναφέροντε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε στην Ιταλία όσον αφορά τους ε, δικαστές αστικού δικαίου. Αυτό έχω να προτείνω. Και ελπίζω να έχω τη συνένεση όλων των βουλευτών, Ιταλών και μη, ώστε να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία μετά από αυτή την ευκαιρία που είχαμε να συναντήσουμε τους ειρηνοδίκες από την Ιταλία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας ε, βοηθάτε τόσο τώρα που θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Κύριε Μπέκερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εφτά παρόμοιες αναφορές έχουμε εδώ. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε μεγάλο όγκο πληροφοριών Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αμοιβέ τους. Κάθε λεπτομέρεια των ε, καθηκόντων των ειρηνοδίκων υπάρχουν. Επίσης το ότι οι ειρηνοδίκες δεν είναι βοηθητικό προσωπικό, ότι σε τακτική βάση ε, ασκούν αυτό το λειτουργήμα. Δύο ερωτήσεις λοιπόν έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι πληροφορίες σας λείπουν και δεύτερον, πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτό. Δεν μπορούν οι αναφέροντες πια να περιμένουν. Φυσικά θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ. Κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ έχουμε μια κλασική περίπτωση παραβίασης της γνωστής ε, συμφωνίας πλαίσιο της 18ης Μαρτίου του 1999 που λέει ότι απαγορεύεται η κατάχρηση και η καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγει ο εργοδότης να συνάπτει συμβάσεις αορίστου χρόνου. Δηλαδή οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες πρέπει να εκπληρώνονται από τους εργαζόμενους με μόνιμες συνθήκες, με διαδικασίες μονιμοποίησης αν είναι στο δημόσιο ή με διαδικασίες αορίστου χρόνου εάν είναι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το ξέρουμε και ισχύει παντού. Όμως όλα τα κράτη-μέλη παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία πλαίσιο. Έχουμε παράδειγμα στην Ελλάδα και έκανα πρόσφατα μία ερώτηση για την μονιμοποίηση αυτών που ονομάζουμε εμείς αναπληρωτές καθηγητές. Και ενώ υπάρχει για το θέμα αυτό και απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα αρνούνται να μονιμοποιήσουν τους αναπληρωτές καθηγητές, οι οποίοι κάνουν την ίδια δουλειά με τους καθηγητές τους υπόλοιπους στα γυμνάσια ή στα λύκεια ή στα σχολεία και όμως δεν μονιμοποιούνται. Εδώ, στην περίπτωση των ε, αναφερόντων έχουμε επίτιμους λέει δικαστές ή ειρηνοδίκες αλλά στην πράξη αποδεικνύεται και το έχουν δεχτεί όλοι το δέχεται και το Ιταλικό Δημόσιο το δέχτηκε η Κομισιόν ότι έχουμε μια καραμπινάτη παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο. Δηλαδή παραβιάζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εφόσον παραβιάζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, η Κομισιόν έπρεπε ήδη να έχει φέρει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση και αυτό είναι συγκεκριμένο. Και δεύτερον, η Ιταλική κυβέρνηση και το Ιταλικό Κοινοβούλιο πρέπει να βρει εδώ και τώρα μία άμεση λύση στο πρόβλημα όλων των αναφερόντων οι οποίοι είναι εδώ, οι οποίοι μας εξέθεσαν τα ζητήματα. Άρα λοιπόν καθυστέρηση δεν χωρά. Εάν λάβουμε υπόψη αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Ιταλικής κυβέρνησης, σημαίνει ότι μέχρι το Μάιο πρέπει να υπάρχει νομοθέτηση και ρύθμιση του ζητήματος. Επομένως, πρώτον, εμείς θέλουμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά, Δεύτερον, να ασκηθεί πίεση και νομίζω ότι από την Ιταλική πλευρά, αν το εννοούν, πρέπει να λύσουν το θέμα. Μην φτάσουμε σε ένα σημείο και πούν, ξέρετε, διαλύθηκε το κοινοβούλιο και θα κάνουμε εκλογέ και θα σα λύσουμε το θέμα στον αιώνα τον άπαντα. Δηλαδή ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν και η Κομισιόν πρέπει να ξεκινήσει τις διαδικασίες επί παραβάση. Να στείλει την επιστολή και από εκεί και πέρα να αρχίσουν να τρέχουν τα δικαιώματα των αναφερόντων, διότι υπάρχει και δικαίωμά τους, και το ξέρουν αφού είναι δικαστές, αποζημιώσεως Εφόσον παραβιάζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωσή τους δικαιούνται να αποζημιωθούν. Να λυθεί λοιπόν το θέμα τους, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς στην Επιτροπή και στηρίζουμε την προσπάθεια των αναφερόντων και ελπίζουμε ότι θα λυθεί το θέμα αυτό. Αλλιώς θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Let me colleagues just point out that we have one... Να αναφέρω συναδελφοί ότι έχουμε άλλη μία αναφορά, οπότε παρακαλώ όταν παίρνετε τον λόγο περιοριστείτε σας παρακαλώ χρονικά στο ένα λεπτό από τώρα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Ελεονόρα, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, προσπαθήστε να είστε πολύ σύντομοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο συνάδελφος κ. Μαριάς. Να επαναλάβω απλά ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων έδωσε μια σαφή ένδειξη για το πόσο σημαντική είναι λειτουργικά οι ειρηνοδίκες ε, σε σχέση με τους ε, ένιστους ε, δικαστές. Όχι μόνο επαναλαμβάνω, αλλά υπενθυμίζω, αναφέρθηκε επίσης, να υπενθυμίσουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2012 επί του θέματος αυτού. η κυβερνητική παρέμβαση με την καταεξουσιοδότηση κατα νομοθεσία του 2016 ουσιαστικά επιδεινώθηκε η κατάσταση. Έγινε ακόμα πιο βέβαιη η κατάσταση των ανθρώπων αυτών. Παγιώθηκε η αβεβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Συμφωνώ λοιπόν με το όσο είπαν οι συνάδελφοι. Ας γράψουμε μια επιστολή, αλλά κυρίως ε, ας ε, διατηρήσουμε την προσοχή μας. Φυσικά ε, πρόκειται για παραβίαση τις νομοθεσίες, οπότε θα ήθελα γρήγορες και σοβαρές ε, παρεμβάσεις στο συντομότερο δυνατόν στο μέτωπο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πολιέζε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος αντικαθιστώ τον κύριο Τσίριο που ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό αλλά που χρειάστηκε να βρίσκεται στην Ιταλία για άλλε δεσμεύσει που είχε. Εγώ έχω παρακολουθήσει την υπόθεση εδώ και χρόνια. Έχω ε, υποβάλει και εγώ κοινοβουλευτικό ερώτημα. Συμφωνώ με τι επικρίσει ε, και την προβληματική που ακούσαμε από αυτή την κατηγορία επαγγελματιών που επαναλαμβάνω ε, ε, διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στο δικαστικό σύστημα της Ιταλίας και η κατάστασή τους αποτελεί παράδοξο από κάθε άποψη αμοιβή, προστασίας, αβεβαιότητας ε, παραβιάζει εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τις άδειες, τις αδεισμητρότητας τίποτα δεν είναι σαφέ ε, για του επαγγελματίε. Οπότε συμφωνώ με τον κύριο Κοτσολίνο, είναι απαραίτητο να παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά και σα. συγχαίρω ε, συγχαίρω και του μη συναδέλφου για την ευαισθησία που δείχνουν. Σα ευχαριστούμε. Είναι ε, μια μάχη πολιτισμού που πρέπει να, ε, φέρει, να καταλήξει ο τέλο το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ιδιαίτερο. Τελευταίο ομιλητή είναι ο κύριο Τέρι Κάμπρα. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομο και μετά θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες. Στην πραγματικότητα... Ε, ουσιαστικά είστε επίτιμοι δικαστές χωρίς λεφτά και χωρίς δικαιώματα. Είναι τρομακτικό αυτό που σας συμβαίνει. Είναι απαράδεκτο. Και το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι και πολύ δύσκολο να επιληθεί. Είναι παλιό και πολύ σημαντικό είναι επίγον και πρέπει να πω έχω μείνει άφωνος μετά όσα άκουσα εδώ. Λέμε ότι θα επιληθεί μέχρι την προθεσμία του Μαΐου. Ναι, ενδεχομένω και μετά η Κομισιόν μας λέει ότι ελπίζει να καταλήξει σύντομα σε μια καλή λύση. Ναι, ξέρετε, άμεσα χρειάζεται η λύση. 20 χρόνια είχατε. Οπότε δεν νομίζω θα σε δύο μήνες θα τα καταφέρετε πρέπει να επιληθεί άμεσα και φυσικά η αναφορά πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα στραφούμε στους δύο αναφέροντες που ήρθαν εδώ αλλά δεν πήραν τον λόγο. Η Παύλα Μαρκέτα. Μπορείτε να είστε πολύ σύντομοι σας παρακαλώ. Το πολύ δύο λεπτά ή και πιο σύντομοι αν μπορείτε και μετά ο Άλμπερτο Ρώση. Αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, Αναφέρομαι στην αναφορά 177 του 2016 για να τονίσω τις πτυχές της ασυμβατότητες. Εδώ και 25 χρόνια οι ειρηνοδίκες ως θεσμός αποτελούν σταθερό θεσμό του Ιταλικού δικαστικού συστήματος όμοιου με τον επαγγελματία δικαστή όπως λέγεται. Ε, επιτελεί λειτουργίες παρόμοιες στο άρθρο 1 του διατάγματος 12 του 1941 για το δικαστικό κανονισμό προβλέπεται ότι ο ειρηνοδίκης είναι έμιστος, τακτικός δικαστής, ανήκει στο δικαστικό σώμα όπως θεσπίζεται από το νόμο 364 του 1991. από τα κοινά χαρακτηριστικά των δύο αυτών δικαστών του τακτικού επαγγελματία και του επίτιμου παρατηρούμε ασυμβατότητα στο θέμα της αμοιβή. Αντιμετωπίζεται διαφορετικά ο ειρηνοδίκης, ενώ οι λειτουργίες του δεν του επιτρέπουν να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρωτεύουσα δευτερεύουσα δραστηριότητα στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε πολιτική ιδιότητα, όπως επιτρέπεται ε, σε μόνιμους δικαστές ε, να αναλάβουν άλλους ρόλους. Ναι, ο Ερηνοδίκης μπορεί να ασκήσει το δικηγορικό επάγγελμα, αλλά λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας είναι αδύνατη η άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. για να καταλάβετε πόσο αδύνατο είναι να ασκήσει οποιαδήποτε ε, εργασία του απαγορεύεται να ασκήσει οτιδήποτε θα μπορεί να υπονομεύσει την εργασία του. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ασκήσει ε, εμπορική δραστηριότητα. Ο Ειρηνοδίκης συμπερασματικά βρίσκεται σε αβέβαιη εργασιακή κατάσταση ενώ αντιμετωπίζεται πιο αυστηρά σε σχέση με τους επαγγελματίες δικαστές όσον αφορά τα καθήκοντά του. Το δικαστικό καθεστώς και η ανανέωση των λειτουργιών του από τα 15 στα 20 χρόνια έρχονται σε αντίθεση με την έννοια της αβεβαιότητας. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, αλλά πραγματικά τα ακούσαμε όλα αυτά ήδη. Δεν έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει λόγος να τα επαναλάβουμε. Ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με την επόμενη αναφορά αξιοπρεπώς πριν κλείσει ο χρόνος και φύγουν οι διερμηνείς. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και να δώσω το λόγο αμέσως στον Αλπεντορόση Κοιτάξτε, θα είμαι πολύ γρήγορος. Εδώ η Ιταλική κυβέρνηση ψεύδεται. Δεν λέει τίποτα άλλο από ψέματα. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή ένας κατεξουσιοδότης νόμος θέλει πραγματικά να κόψει τα πόδια των επίτιμων δικαστών δικαστές που εργάζονται με πλήρες ωράριο και αυτή η εξουσιοδότηση νομοθεσία θα μετατρέψει την εργασία πλήρους απασχόλησης σε εργασία μερικής απασχόλησης. Θέλει ουσιαστικά να περικοπούν οι αμοιβέ μας και η κοινωνική μας ασφάλεια να μειωθεί. Δηλαδή η διακριτική μεταχείριση δική μας. Μας κοροϊδεύουν μου κάνει έκπληξη αυτό που είπατε κύριε Κοτσολίνα. Το πρόβλημα δεν είναι να εφαρμοστεί η νομοθεσία, η κατεξοδότηση νομοθεσία μέχρι το Μάιο, αλλά να καταργηθεί, διότι πρόκειται για προσβολή ε, προς την ανεξαρτησία των δικαστών και τα δικαιώματα των 5.000 οικογενειών ε, που βασίζονται σε αυτή την εργασία εδώ και μια 20 ετία. Ουσιαστικά μας κοροϊδεύουν. Θέλουμε αμέσως να αποσυρθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία επί κατά της Ιταλικής κυβέρνησης η οποία το μόνο που προσπαθεί είναι να κερδίσει χρόνο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί καμία από τις παραβιάσεις αυτές. Αυτή είναι η αλήθεια, αξιότιμε κύριε. Αν θέλετε να το σημειώσετε, ωραία. Αλλιώς ε, μπορούμε να προχωρήσουμε και επάπειρον, χάνοντας ε, χρόνο, διότι εδώ μας κοροϊδεύουν. Άνθρωποι πεθαίνουν, ξέρετε κύριε. Υπάρχουν συνάδελφοι που μία εβδομάδα μετά, επειδή δεν είχαν δικαίωμα άδεια ασθενεία, πέθαναν στο δικαστήριο μέσα. Υπάρχουν συνάδελφοι που πάνε να δουλέψουν ε, εκτός έδρας έχουν κάποιο ατύχημα μένουν παράλυτοι, χάνουν τη δουλειά τους και η Ιταλική κυβέρνηση δεν τους αναγνωρίζει καν την υπηρεσία τους. Είναι ντροπή κύριοι, είναι ντροπή το να υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές που λένε ότι θα περιμένουμε μέχρι το Μάιο, να περιμένουμε τι, ε, μια κατεξουσιοδότηση νομοθεσία που θέλει να μας ακυρώσει, να μας καταργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω μας εξηγήσατε πολύ καλά την υπόθεσή σας και είναι μια από τις στιγμές που είμαι περήφανη που είμαι πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, διότι υπάρχει ομόφωνη υποστήριξη ε, από όλους τους συναδέρφους, από όλες τις διαφορετικές πολιτικές ομάδες σχετικά με το πώς θα προχωρήσουμε. Θα παραμείνει ανοιχτή αναφορά και θα την ε, απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κύριε ε, παραθέτω τα λόγια σας τι παραπάνω πληροφορίες χρειάζεστε και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα πρώτου να αναλάβετε δράση. Και θα στραφούμε και στην ε, Ιταλική Επιτροπή Αναφορών, όπως ε, ανέφερε ο συνάδελφος ε, Κωνσταντίνο, για να έχουμε περαιτέρω διάλογο μαζί τους και θα στείλουμε μια πολύ ακριβή επιστολή ε, στον ε, Υπουργό Δικαιοσύνη της Ιταλίας και θα το ρωτήσω η κυβέρνηση της Ιταλίας πώς θα λύσει την κατάσταση και πώς θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα της Ιταλίας, διότι αυτό διακυβεύεται εδώ. Θα εκμεταλλευτούμε λοιπόν την ορμή που έχει δοθεί στο θέμα αυτό και θα καταστήσουμε το θέμα αυτό απόλυτα σαφές. Επίσης θα αναφέρουμε αυτό που είπατε εσείς, ε, τον αριθμό των οικογενειών δηλαδή, που επηρεάζονται από αυτήν την πολύ περίεργη κατάσταση και κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε. Χρειάζεται αναγνώριση αυτής της κατηγορίας ε, δικαστών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, βλέπω όλοι να αντιδρούν θετικά. Ε, απευθύνομαι λοιπόν σε εσά, ε, κύριοι αναφέροντε, ε, να μείνετε ήσυχοι. Παίρνουμε απολύτω στα σοβαρά την αναφορά σα και θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες πάνω στο θέμα αυτό. καλή επιστροφή λοιπόν στην Ιταλία και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να λυθεί το πρόβλημά σας. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο για την επόμενη αναφορά και ζητώ συγγνώμη από τους αναφέροντες για το θέμα αυτό. Είναι η αναφορά 429 ε, σχετικά με ε, το ε, έργο αστικοποίησης στην Βαλένθια, στη Σκαλαμόσκα. Και έχουμε εδώ τους αναφέροντες, Ρόμπερτ Χιουλίστον, και Μάρτα Γιουλέν ε, και θα μοιράσετε το χρόνο μεταξύ σας. Ε, κύριε Χιουλιστόν, έχετε το λόγο πρώτος. Παρακαλώ. Παρακαλούμε όσους αποχωρούν από την αίθουσα να το κάνουν ε, σύντομα και πολύ ήσυχα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εμείς στην επόμενη αναφορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε πολύ ευγνώμονες στην Επιτροπή Αναφορών που ε, κράτησε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη από τότε που υπευλήθη η αρχική αναφορά το 2010 με την υποστήριξη 7.000 υπογραφών. Εφτά χρόνια μετά κυρία Πρόεδρε, φτάσαμε σε μια αποφασιστική στιγμή για τον καθορισμό του μέλλοντος του τελευταίου αυτού χιλιόμετρου σε γη στην Οριγουέλα Κώστα. Τα άλλα 15 χιλιόμετρα έχουν οικοδομηθεί τελείω μέχρι, την, ε, μέχρι τη θάλασσα. Και έχει αναζωογονηθεί η αγορά ακινήτων σε αυτό το μέρος της Ισπανίας ε, και ε, ο οικονομικός φορέας ε, στόχο έχει να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του να αναγύρει 1.500 νέες κατοικίες καθυστέρησαν ε, και παρέλυσαν τα σχέδια του ε, λόγω της επιμονής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, του, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, διενεργηθεί μελέτη αντικτύπου, περιβαλλοντικού αντικτύπου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2014 από τον ίδιο τον ανάδοχο, το οποίο όμως δείχνει σύγκρουση συμφερόντων. Η μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, επικρίθηκε ευρέως ε, όταν δημοσιεύθηκε. Το δικό μας ε, μικρό πολιτικό κόμμα υπέβαλε 7.500 αντιρρήσεις. Οι πιο σημαντικές αντιρρήσεις όμως προέρχονταν από τους υπαλλήλους, τους αρμόδιους για το περιβάλλον στο Δημαρχείο της Ορυχοέλα δεν προστατεύονται δύο απειλούμενα είδη στην Καλαμόσκα, ένα σπάνιο φυτό και ένα σπάνιο σαλιγκάρι και ε, επέκριναν τις προτάσεις ε, διότι δεν σέβονται τα όρια οικοδόμησης και δεν λαμβάνουν υπόψη δεν σέβονται τα δικαιώματα των ε, ζώων και επίσης επέκριναν ε, τον κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο αυτού του έργου. Επίσης ακούστηκαν επικρίσεις ε, που δεν ε, λήφθη υπόψη η διαθεσιμότητα νερού εάν αυξηθεί ο πληθυσμός της Καλαμόσκα κατά 20%. Το 2014 δεν είχαμε σημαντικές τροποποιήσεις κυρία Πρόεδρε. Οι πολίτες και οι κάτοικοι αγωνίζονται σε έναν άνισο αγώνα, διότι ο ανάδοχος είναι μια επιχείρηση οικοδομών ε, με πολύ επιρροή και με πολύ κεφάλαιο μπορεί να αγοράσει την επιρογνωσία που χρειάζεται και οι τοπικές αρχές βρίσκονται υπό Πολύ πίεση. Ε, καλούμε λοιπόν την Επιτροπή Αναφορών να ε, δημιουργήσει συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκίλεν. Θα έχει να προσθέσει κάτι ή να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να αρθρώσουμε εδώ μια διεκδίκηση που έχει να κάνει με τη δική μας επικράτεια γιατί το τελευταίο ελεύθερο χιλιόμετρο παραλίας απειλείται από την κατασκευή 1500 κατοικιών. Έγινε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων χάρη στην Επιτροπή σας η οποία μελέτη όμως εξαπατά. Υποτίθεται ότι επί χάρτου φαίνεται ότι πληρούνται οι διατάξεις που είχε προβλέψει η Επιτροπή στο ψήφισμά Ωστόσο η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι αρμόδιες αρχές δεν εξετάζουν το θέμα από όλες τις απόψεις, αγνοούν την ύπαρξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε περίπτωση προς, ε, καθορίζεται ένα, προστα... ένα σχέδιο προστασίας του ε, Αιγιαλού που δεν περιλαμβάνει την προστασία αυτής της ζώνης ενώ είναι απολύτως απαραίτητη ε, να... η προστασία αυτής της ζώνης. Ζούμε σε μια χώρα όπου τελικά είναι αδύνατο να αντιταχθεί κανείς στα πολεοδομικά σχέδια παρόλο που καταστρέφονται μοναδικά οικοσυστήματα όπως το συγκεκριμένο και παρόλο που ε, καταδικάζονται οι άνθρωποι να ζουν σε κοινότητες ε, ε, με απερίμωση, με συνθήκες απερίμωσης, χωρίς επαρκείς δημόσιες υπηρεσίες και με μαζική συσσόρευση, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο το οποίο έχει πληγώσει ανεπανόρθωτα την επικράτειά μας. Στην Οριγουέλα είναι πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι από όλα τα μετερίζια που έχουν ενωθεί σε αυτή τη διεκδίκηση. Είναι κόσμος που ελπίζει στην Ευρώπη, που δεν θέλει να χάσει τις ελπίδες του σε αυτήν ε, για αυτό το έργο το οποίο βρίσκει αντίπαλη και αντίθετη όλη την τοπική κοινωνία στο σύνολό της η οποία σύσσωμη αντιτάσσεται σε αυτό το έργο. Ε, είναι μια τεράστια πρόκληση για να δούμε τι είδους κοινωνία και τι είδους κοινωνικό μοντέλο θέλουμε στο, ε, στο τέλος για το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ο Ράμος Φλωρέδο, εκπρόσωπος της Επιτροπής, είναι εδώ. Παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Δεν υπάρχει χρόνος πράγματι και την αναφορά αυτή την έχει συζητήσει η Επιτροπή σας το 12 και το 14. Επομένως θα επαναλάβω τη γραπτή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα υπενθυμίσω ότι χάρη στην παρέμβαση της Επιτροπής Αναφορών και στην αναφορά σας και χάρη στην ε, υπόθεση που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτή την αναφορά, οι αρμόδιες ισπανικές αρχές, ο Δήμος και η αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια άλλαξαν το αρχικό του σχέδιο όπου θεωρούσαν ότι δεν εφαρμόζεται η οδηγία για την ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό ήταν που δεν δεχόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το συμμορφώθηκαν οι Ισπανικές αρχές. Πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία, πρέπει να γίνει εξέταση, πρέπει να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το παράρτημα 2 της ε, οδηγίας και μετά από το screening, από αυτή την εξέταση, ε, βασικό συμπέρασμα είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να ρυθμιστεί περιβαλλοντικά πριν δοθούν άδειες χορηγήσεις, εγκρίσεις και το καθεξής. Ε, με τις διαθέσιμες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι Ισπανικές αρχές δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επομένως δεν έχει ενδείξεις για να θεωρεί ότι οι Ισπανικές αρχές δεν θα το πράξουν και δεν θα εφαρμόσουν αυστηρά το κοινοτικό περιβαλλοντικό δίκαιο και δηλαδή την οδηγία αξιολόγηση περιβαλλοντικού Λαμβάνοντα αντικτύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές αξίες της περιοχής. Θα ήθελα να πω ότι βασικός στόχος της οδηγίας αυτής είναι η προστασία του περιβάλλοντος, όμως είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνονται. Πρώτον, συγκεκριμένη και επίσημη διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι εκάστοτε εθνικές αρχές και δεύτερον, συμμετοχή του κοινού, συμμετοχή της κοινωνίας και άρα οι δημόσιες αρχές τίθενται ενώπιον των ευθυνών τους με διαφάνεια έναντι στην κοινωνία. Ελπίζουμε και περιμένουμε να τηρηθεί ε, απαρέγκλητα η διαδικασία η περιβαλλοντική. Είναι δεσμευτική η γνωμοδότηση σύμφωνα με, με την Ισπανική νομοθεσία και άρα θα μπορούν οι Ισπανικές αρχές να λάβουν την πιο κατάλληλη απόφαση σε σχέση με αυτό το έργο. Ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε ακόμα τρεις ομιλητές στον κατάλογο. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ε, να κινηθούμε όπως με την προηγούμενη, δηλαδή με μεγάλη συνένεση. Οπότε μην ε, μιλήσετε πολύ παρακαλώ. Ευχαριστώ να σας πω ότι όλες οι αναφορές είναι το ίδιο σημαντικές και όλες αξίζουν να αντιμετωπιστούν με το σωστό τρόπο. Δεν είναι δίκαιο κάποιες αναφορές να τις εξετάζουμε μισή ώρα και άλλες μόνο δέκα λεπτά. Εάν τώρα ε, θεωρείται ότι δεν έχει συζητηθεί σωστά, να τους ξανακαλέσουμε τους αναφέροντες και να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση με ε, σωστές ε, προϋποθέσεις και όχι να έχουμε ένα λεπτό μόνο ο καθένας. Τούτων λεχθέντων, να ευχαριστήσω τους αναφέροντες για τον αγώνα που δίνουν, που κάνουν. Να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η απάντηση που αναφέρατε είναι απάντηση γραπτή του 2012 Πώς είναι δυνατόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναλαμβάνετε και να αναμασάτε πράγματα του 12. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια, ένα σωρό πράγματα έχουν παρευληθεί. Δεν μπορείτε να μας παραπέμπετε στην αγραπτή σας απάντηση του 12 θα περίμενε κανείς να έχει γίνει αξιολόγηση του θέματος, εξέταση και να έχετε μια απάντηση επί της ουσίας, κατάλληλη, επαρκής, που να ανέρχεται στο ύψος των περιστάσεων. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Αυτή η αναφορά μας έρχεται για την αυτόνομη ε, κοινότητα της Βαλενθία, για το Ισπανικό κράτος, οικιστικές ε, καταχρήσεις, απειλή για το τοπίο, για το φυσικό τοπίο, για το περιβάλλον. Είναι η τελευταία γωνιά ελεύθερης παραλίας σε μια ολόκληρη περιοχή. Έχουμε δεκάδες χιλιόμετρα ε, αιγιαλού ε, που έχουν χτιστεί, που είναι δομημένα και έχουμε ένα μόνο τελευταίο χιλιόμετρο ελεύθερης γης, ελεύθερου αιγιαλού. Ε, και ε, συζητούμε ξανά και ξανά για τη φούσκα των ακινήτων, για το πώς δεν θα ξανασυμβούν τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να ασχοληθούμε με το περιβάλλον, να το προστατεύσουμε και να το σεβαστούμε. Υπ' αυτή την έννοια. Η Επιτροπή μας ζητήθηκε να υπάρξει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν περιλαμβάνει τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο για, ε- την παράκτια ζώνη, για τον Αιγυαλό ε- ε- και δεν περιλαμβάνει και ε, το ότι δύο προστατευόμενα είδη υπάρχουν στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Επιτροπή μας όμως πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσο αυτή η μελέτη είναι επαρκής. Μας λένε ότι δεν είναι επαρκής. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό και πολύ σοβαροί. Ως Επιτροπή Αναφορών λοιπόν να απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές, άρα στις αρχές της αυτόνομης κοινότητας της Βαλένθιας, να γίνει ανεξάρτητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι ε, μελέτη που κάνει η ίδια η αυτόνομη κοινότητα η οποία είναι ενδιάδικο και ενδιαφερόμενο μέρος. Να ε, ασχοληθεί η μελέτη με τα προστατευόμενα είδη, με την έλλειψη των, ε, πόρων, ή των υδάτινων πόρων μεταξύ άλλων και να καλέσουμε τις ε, αρχές να προστατεύσουν αυτή τη ζώνη. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να την προστατεύσουμε. Ε, ως Επιτροπή Αναφορών το ε, ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνει σωστά αυτό που ζητήσαμε. Ζητήσαμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν έγινε σωστά. Οφείλουμε να απευθυνθούμε στις αρχές της αυτόνομης κοινότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Κάμπρας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν συζητάμε για πολύ χώρο, μιλάμε για ένα χιλιόμετρο. Αλλά είναι κρίσιμη σημασία. Δεν θα μιλήσω για την ε, μαζική αστικοποίηση την οποία θεωρώ φρικτή. Θα μιλήσω για τα νομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Η περιβαλλοντική μελέτη είναι μεροληπτική. Σε καμία περίπτωση δεν αξιολογήθηκε και δεν αντιπαρατέθηκε με μια επίσημη έκθεση όπως ε, όμως ε, ε, υπάρχει εντολή να γίνει. Άρα δεν έγινε σεβαστή αυτή η εντολή. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λέτε να περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος από το 2012. Εάν το 2012 παραμείνει, λοιπόν, παρέμεινε λοιπόν ανοιχτή η αναφορά, ε, τότε πρέπει να παραμείνει και τώρα. Γιατί δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή και καμία πρόοδος. Αυτή είναι η γνώμη μου λοιπόν. Πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ευχαριστώ η Ρώσα. Ε, συντομία κυρία Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει πράγματι να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Οι αρχές της Βαλένθια θα πρέπει να απαντήσουν. Στις 27 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η εξέταση του θέματος η δημόσια, θα καθαρογραφεί η συζήτηση και εγώ έχω εμπιστοσύνη στις Ισπανικές αρχές, είναι ανεξάρτητα τα όργανα της Γενικής Διεύθυνσης, άλλωστε είναι η αριστερά στην εξουσία στην αυτόνομη αυτή κοινότητα, αλλά εν πάση δεν έχει σημασία η πολιτική χρειά. Οι εκθέσεις πάντοτε συντάσσονται ανεξάρτητα. Τα δικά σας κόμματα, οι δικές σας πολιτικές ομάδες είναι στην εξουσία, τεωρικά και Αλβιόλ. Νομίζω ότι η έκθεση θα είναι πολύ ενδελεχή. Θα ζητήσουμε αυτό, να τηρηθεί η νομοθεσία, να γίνουν τα δέοντα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Είμαστε σε θέση να κλείσουμε αυτή την αναφορά με τρόπο που θα ε, συμφωνήσουν οι αναφέροντες και θα αποφύγουμε πολύ μεγάλη επιθετικότητα από άλλους συναδέλφους. Επομένως, πρώτον, κρατούμε την αναφορά ανοιχτή. Δεύτερον, στέλνουμε επιστολή στις αρμόδιες αρχές και λέμε ότι αυτή, η αναφορά ενδιαφέρει την Επιτροπή μας πάρα πολύ ε, τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια και βασιζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Άρα να αξιολογήσει την αξιολόγηση αντικτύπου που έγινε έγινε Αυτό είναι το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απάντηση γραπτή. Αυτό θα ήταν εξαιρετικό. Και στην επιστολή θα τονίσουμε ότι βεβαίως η οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως, απολύτως και ότι μας ανησυχεί ιδιαίτερως αυτή η ζώνη, παρόλο που δεν είναι μεγάλη έκταση, είναι εξαιρετικά ευαίσθητη έκταση ένα ευαίσθητο και όμορφο τμήμα της ευρωπαϊκής επικράτειας. Θα επανέλθουμε λοιπόν και έτσι θα πράξουμε και θα συμπεριλάβουμε το σημείο στην ημερήσια διάταξη μόλις υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι οι αναφέροντες είναι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι μπορώ να σας ευχηθώ καλή επιστροφή. Και ένα λεπτό για την έκθεση της διερευνητικής αποστολής στη Σουηδία και με αυτά θα ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστώ τους αναφέροντες τους χαιρετώ. Ε, δίνω το λόγο στον αρμόδιο για το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματοποίησαμε λοιπόν ερευνητική επίσκεψη πέρσι στη Σουηδία. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις με τις Σουηδικές Αρχές πολύ ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις. Και προσωπικά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει σαφής βούληση από τις αρχές της Νότιας Σουηδίας να λύσουν το πρόβλημα και θα ετοιμάσουμε την ε, έκθεσή μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πάλι που ήσουν τόσο τόσο ε, υπομονετικός και ε, ευγενικό κατά τη διάρκεια τη επίσκεψη αυτή. Ευχαριστώ και όλου του Γερμηνεί, λέει η και εμεί ευχαριστούμε και καλή όρεξη. Καλό βραδινό. Σα ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Θα τα πούμε σύντομα.